Το σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη ότι δεν υπάρχει διαδικασία catch the eye για αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σεφκοβιτς, εξ ονόματος της Επιτροπής. Vice President Sefcovic, you have the floor. Με μεγάλη χαρά είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013 που μόλις υιοθετήθηκε από το σύνολο των Επιτρόπων. Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει τον εντατικό πολιτικό διάλογο και συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και με τη διάσκεψη των Προέδρων και ο διαρθρωμένος διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις επιμέρους κοινοβουλευτικές επιτροπές ήταν πολύ βαθύτερος από ό,τι πέρυσι. και είχαμε και τις τελευταίες πρόσφατες ανταλλαγές απόψεων με την διάσκεψη των Προέδρων, στην οποία συμμετείχα και εγώ συλλέξαμε πληροφορίες οι οποίες μας χρησιμεύσαν για τη διαμόρφωση του προγράμματος εργασίας. Μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάναμε προσπαθούμε να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί στις πιο βασικές θα έλεγα προτεραιότητές μας που είναι η ανάπτυξη, η επιστροφή στην ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η αντιμετώπιση της κρίσης και η πορεία προς την βιώσιμη και φόρο ανάπτυξη. Και μετά από αυτά που ακούσαμε το πρωί μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα φάρμακο και ότι όλα τα επίπεδα της κοινωνίας θα πρέπει να πάρουν μέρος στην προσπάθεια. Να δούμε πώς λοιπόν και το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συνεισφέρει και πως η προσπάθεια αυτή είναι κάτι το οποίο θα προσελκύσει και το εκλογικό σώμα το 2014. Εφτά είναι οι βασικές πολιτικές. Πρώτον, να προχωρήσουμε προς την πραγματική Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Εδώ είναι σαφές ότι η πορεία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε μια ενότητα πολιτική και δημοκρατική. Δεύτερον, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, όθηση στην ανταγωνιστικότητα. Τρίτον, δημιουργία δικτύων στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη. Τέσσερα είναι η ανάπτυξη για τη θέση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά κατηγοριών όπως των νέων σαν παράδειγμα. Θα πρέπει επίσης πέμπτο, να χρησιμοποιήσουμε σωστά τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκτον να δώσουμε το αίσθημα ασφάλειας, ένα δίκτυο ασφαλείας στους πολίτες και τέλος να ενισχυθεί γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν παγκόσμιος παίκτης. Το πρόγραμμα εργασίας λοιπόν σαφώς και περιγράφει και σχεδιάζει τους στόχους, δείχνει το τι ελείπει σήμερα και περιγράφει και τους τρόπους τους οποίους θα ακολουθήσει η Επιτροπή. Να μου επιτρέψετε να σταθώ σε κάποιες από τις βασικές προτεραιότητες. Η δημιουργία, η προσπάθεια μιας πραγματικής και γνήσιας Ευρωπαϊκής και Νομισματικής Ένωσης βρίσκεται στο κέντρο της προσπάθειας. Όπως έδειξε η συζήτηση σήμερα το πρωί, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα ένα πρόγραμμα το οποίο θα προσπαθήσει να συνεισφέρει στη συζήτηση που ξεκίνησε. Προσπαθούμε να είμαστε φιλόδοξοι επί τη βάση των διαθεσίμων μέσων για να διασφαλίσουμε πλήρη δημοκρατικό έλεγχο. Το να το πετύχουμε αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να εξυγχρονίσουμε τους τρόπους με τους οποίους ε, παράγουμε δημόσια έσοδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανταποκριθεί στο αιτήματα των κρατών μελών που θέλουν να προχωρήσουν γρήγορα με τον φόρο για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις διευκολύνουμε. Ο καθένας λοιπόν εδώ θα αναλάβει το μερίδιο ευθύνης και προσπάθειας που του αναλογεί. Έτσι περιμένουμε και από τον χρηματοοικονομικό τομέα να βοηθήσει να αναπτυχθεί η οικονομία με πραγματικούς όρους το 2013 θα ασχοληθούμε με τα θέματα των σκιωδών τραπεζικών δραστηριοτήτων. Οι επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες περιουσιών δεν μπορεί να είναι ευάλωτοι σε ε, καταστάσεις ανεξέλεγκτες. Προσπαθούμε να αλλάξουμε με νομοθετικά πρώτα μέτρα τον έλεγχο και την εποπτεία των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και των αγορών θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Η σταθερότητα είναι η βάση για την σωστή ανάπτυξη. Η εμπειρογνωμοσύνη και η εμπιστοσύνη είναι τα βασικά μέσα εμείς μπορούμε να επιβιώσουμε με μια ιδιαίτερα εξυγχρονισμένη βιομηχανική βάση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε μια ισχυρή ενιαία αγορά, χρειάζεται να καλύψουμε τα διακανονιστικά κένα και να ολοκληρώσουμε την λεγόμενη ψηφιακή οικονομία, να βελτιώσουμε την κινητικότητα ε, σαν κινητήρα και για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές. Είδατε ποιε είναι οι προτάσει της Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ενιαία αγορά. Θα πρέπει οι δράσεις αυτές να εφαρμοστούν εφόσον συμφωνηθούν πριν από το 2014. Η συμφωνία για το πακέτο FMI, δηλαδή για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι κάτι το οποίο είναι προϋπόθεση και εφόσον συμφωνήσουμε εκεί θα μπορέσουμε να στρέψουμε την προσοχή μας και τις προσπάθειές μας του χρόνου στην ολοκλήρωση των τομεακών μέσων και προγραμμάτων. Το 2013 θα ξεκινήσουν και νέες πρωτοβουλίες για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη μείωση του κόστου σε τομείς όπως το ΦΠΑ, τις μοχλεύσεις σε διάφορους τομείς όπως φαρμακευτική βιομηχανία, αεροναυτική βιομηχανία κτλ. Απαιτείται επίσης να δώσουμε μακροπρόθεσμη βεβαιότητα και αίσθηση εμπιστοσύνη στους επενδυτές. Η ε, ε, βελτίωση των υποδομών και στον τομέα της πληροφορικής είναι κάτι το απαραίτητο για να το πετύχουμε τους στόχους που ανέφερα. Όλοι αυτοί είναι λόγοι επίσης για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας και με τον ιδιωτικό τομέα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε την Ευρώπη πρέπει να βασιστούμε στους νέους. Η κρίση των, της ανεργίας των νέων είναι μια κρίση μέσα στην κρίση. Είναι μια κρίση η οποία έχει βάλει στο περιθώριο μια ολόκληρη γενιά και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε σαν κοινωνία και αν πολλοί από τους παίκτες στην περίπτωση και τη μοχλή δράση είναι εθνική και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κινητικότητα, με την βελτίωση της κατάρτισης μπορούμε να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην δημιουργία για να έρθουμε κοντά στην δημιουργία μιας λεγόμενης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας σε συνεργασία με όλους και τον Δεκέμβριο προτείνουμε, θα προτείνουμε και ένα πακέτο για την απασχόληση και το θέμα των εγγυήσεων για την απασχόληση των νέων. Είμαστε αγαπητά μέλη μια κοινότητα αξιών και δεν θα πρέπει όμως να αγνοούμε την οικονομία που είναι ο κύριος παράγοντας των δραστηριοτήτων μας. Για να αναπτυχθούμε και να αναπτύξουμε ε, αριθμούς μεγάλους θέσεων απασχόλησης πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να προστατεύσουμε τους πολίτες. Συγκεκριμένες δράσεις απαιτούνται το 2013 για τη βελτίωση της <clears throat> κινητικότητας, τη βελτίωση της συνεργασίας σε πολλούς τομείς, έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να ασκούν τη δραστηριότητέ τους με ένα αίσθημα ασφάλειας θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις ευρωπαϊκές αξίες σε όλο τον κόσμο και στο εξωτερικό εμπόριο αυτό είναι κάτι που θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Έχουμε την δυνατότητα για τη δημιουργία 2 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης μεσοπρόθεσμα. Η συνεργασία μας με σημαντικούς εταίρους όπως η Ιαπωνία και η ΙΠΑ θα είναι καθοριστική. Θα πρέπει να παίξουμε ένα θετικό ρόλο παγκόσμια και αυτό το αναγνώρισε άλλωστε και η Επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ για μια πραγματική ανάπτυξη και της ανθρωπιστικής βοήθειας και η πολιτική γειτονία και κυρίως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή και στην περιφέρειά μας αλλά και ακόμα πιο μακριά. Και γι' αυτό δημιουργούνται νέα προγράμματα νέας γενεάς που θα συνεισφέρουν και ως προς αυτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, είναι κρίσιμη η καιρή. Τα βήματα που θα πάρουμε τα επόμενα χρόνια θα αποφασίσουν για το μέλλον μας. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τις δυνατότητές μας έτσι ώστε το υπόλοιπο αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου να είναι παραγωγικό σε σχέση με τις ανάγκες μας για το 2014 και μετά. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρξει πρόοδο σε όλα τα προγράμματα και να πάρουμε τα βήματα που απαιτείται από κοινού για μια ισχυρότερη και πιο ευημερούσα Ευρώπη ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Γιώζεφ Σάζερ, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρωτού εκφωνήσω τον λόγο μου, επιτρέψτε μου, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για την Επανάσταση και τον αγώνα για την ελευθερία του 1956 να υπενθυμίσω κάποια πράγματα στην Ουγγαρία. Ξεκίνησε αυτή η Επανάσταση όπως στη σημερινή μέρα τότε και επί ε, ημέρες η κυβέρνηση της Ουγγαρίας επετίθετο κατά του ιδίου του λαού της. Ήταν πραγματικά κάτι αναξιοπρεπές και πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013 είναι ένα στρατηγικού χαρακτήρα έγγραφο. Το Κοινοβούλιο στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές αλλά και στην Ολομέλεια εξετάζει αυτά τα θέματα επί αρκετό χρονικό διάστημα. Μόνο μπορούμε να ακούσουμε από την περιγραφή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα σχετικά με το νέο φόρο. Αλλά θα ήθελα να καλωσορίσω εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προθυμία να αποδεχθεί κάποια από τα στοιχεία τα οποία συζητήθηκαν εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο στο παρελθόν και που έχουν συμπεριληφθεί και στο ψήφισμά μας του Σεπτεμβρίου. Προφανώς πρέπει να πω ότι σε αυτή την κρίση σε αυτήν την περίοδο έκδηλης κρίσης πρέπει να συνειδητοποιήσουμε περισσότερο τα θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού αλλά θα ήθελα να τονίσουμε και ότι όπως και στο ψήφισμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να, είναι, να δείξουν ευελιξία και να αντιδρούν άμεσα σε διαφορετικές καταστάσεις. Θα ήθελα να παριθμίσω κάποια από τα σημεία που η ομάδα μας, το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θεωρεί ως προϋπόθεση για την υποστήριξη του προγράμματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι προφανές ότι υποστηρίζουμε και υπερασπιζόμαστε το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τις εξουσίες της και τι αρμοδιότητες της υπέρ του προγράμματος αυτού. Είμαστε, ενθαρρύνουμε και θα θέλαμε να δούμε καλύτερη χρήση εντολήν πράξεων, εντεταλμένων πράξεων που και σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να βοηθήσει τον ελεγκτικό ρόλο από πλευράς του Ευρωκοινοβουλίου εναντί του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά προφανώς και εναντί του έργου που επιτελούν και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν είναι πρόθυμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει το επαχθές γραφειοκρατικό βάρος, ρυθμιστικό, κανονιστικό και άλλο βάρος και σε σχέση και με το βάρος της κρίσης να υπάρξει κάποια ανακούφιση Γενικά δεν μπορούμε να ρυθμίζουμε τα πάντα και ο επιπαντός του επιστητού. Η κρίση το έδειξε αυτό. Υπάρχουν ανάγκες για κάποιες ρυθμίσεις, αλλά το συνολικό ρυθμιστικό βάρος ε, που είναι επαχθές πρέπει να μειωθεί. Και επίσης όταν είναι πρόθυμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί στην εφαρμογή, παρακολούθηση εφαρμογής ε, στον ρυθμό και στην ε, ταχύτητα που ακολουθείται, είναι κάτι σημαντικό σε σχέση με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή νομοθετικού έργου, για παράδειγμα. Θα θέλαμε να υποστηρίξουμε την πολιτική φιλοδοξία και το όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση σφαιρικά και συνολικά, ιδιαίτερα σε σχέση με τα όσα εξέθεσε στον λόγο του ο πρόεδρος Μπαρόζο στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου, στον λόγο του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προφανές ότι οι ευρωβουλευτές που άμεσα εκλέγονται ως αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών λογοδοτούμε για τις πράξεις ή παραλήψεις και έτσι λοιπόν ζητούμε, διεκδικούμε την πρόσθετη τη αξία μέσω των δράσεων και είμαστε πρόθυμοι άμεσα να αντιδρούμε σε διαφορετικές καταστάσεις χρησιμοποιώντας μια διεργασία fast track ταχεία ε, ρύθμισης, διευθέτησης ε, οποτεδήποτε χρειάζεται αυτό και είναι επίγον προς, το, προς όφελος των πολιτών αλλά επίσης θα ελέγχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσον αφορά την αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων των φορολογουμένων. Θέλουμε να υποστηρίξουμε επίσης και την γραμμή τη που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον τομέα της πολιτικής συνοχής. Αναφέρατε την ανεργία των νέων που και αυτό μας απασχόλησε ε, τις εχθές και επίσης και την δυνατότητα την, ε, χρήση, της χρήσης, της, την απασχολησιμότητα των υπερηλίκων και υποστήριξη επίσης ε, της κινητικότητας από πλευράς τους. Και αυτό που τόνισε ο Αντιπρόεδρος, να δημιουργηθούν τα αναγκαία μέτρα για να ενισχυθεί, να ενδυναμωθεί η Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο για το κόμμα μας. Προφανώς η πλήρη υλοποίηση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς με ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σημαντικό σημείο και αυτό. Και τελευταία μου παρατήρηση που απορρέει από όλα αυτά, όταν κάνουμε κάτι και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πρέπει να αντανακλά αυτό, θα πρέπει να αφορά ένα οδικό χάρτη, ένα χρονοδιάγραμμα δεσμευτικά, τι θα πρέπει να γίνει του χρόνου το 2013. Αλλά πάλι ε, ταχύτητα στις αντιδράσεις μας και ελαστικότητα, διότι η υπευθυνότητά μας, η ευθύνη μας δεν σταματά στην, ε, στο σχεδιασμό με βελτιώσεων αλλά και τη δημιουργία ενός ε, καινοτόμου πλαισίου ώστε να μπορούμε να αντιδρούμε έγκαιρα στα διάφορα στοιχεία της κρίσης. Με αυτές τις προϋποθέσεις θέλω να δηλώσω ότι υποστηρίζουμε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, And Ευχαριστώ κύριε Σάιερ. Εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής και Δημοκρατικής Ομάδας θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκουερέρο Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Επίσης, σε διάφορε παρεμβάσει σα και στην ομιλία για την κατάσταση τη Ένωση, μα είπε ο κύριο Μπαρόσο πω η κρίση τη ε, ανεργία είναι ένα στοιχείο κλειδί για να λύσουμε το πρόβλημα τη οικονομική κρίση γενικότερα. Και μα είπε πω η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι δίκαιη, γιατί η ανισότητα δεν είναι βιώσιμη. Μας είπε επίσης πως η συνολική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται από το κοινωνικό μοντέλο. Πιστεύω πως έχει κάνει σωστή διάγνωση. Είναι σωστή η διαπίστωσή του, αλλά έχει μείνει στα ωραία λόγια, γιατί μεταξύ των λόγων του κυρίου Μπαρόσο και του κυβερνητικού προγράμματος της Κομισιόν υπάρχει μια αδιάβατη άβυσος. Αν δούμε τώρα τι συνέβη με το πρόγραμμα για το 2012, πάνω από το ίμιση των προγραμμάτων της Κομισιόν δεν τελείωσαν. Για παράδειγμα, για τη στρατηγική για την υγεία, τα δικαιώματα των εργαζομένων, για την σωματική ακυρεότητα, για την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων. Όλα αυτά επηρεάζουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Όπως επίσης και η οδηγία για τον καπνό, που ελπίζω πως σύντομα θα φτάσει να περάσει και από το Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν η Κομισιόν μένει κάτω από τη βάση για το πρόγραμμα του 2012 και απογοητεύει για το 2013. Πού είναι τα μέτρα για να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων. Τι θα μας δώσει η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Πού είναι οι δεσμεύσεις μας για τον κοινωνικό διάλογο. Οι ανεργίες στους νέους στην Ευρώπη είναι πάνω από το 20% και σε κάποιες χώρες πάνω από το 50%. Θέλουμε λοιπόν κάποιες εγγυήσει για την απασχόληση των νέων, αλλά χρειαζόμαστε μια πιο επιθετική στρατηγική που θα έχει γίνει αντικείμενο καλύτερου συντονισμού. Αλλά το χειρότερο στο πρόγραμμα εργασία είναι ότι δεν εμφανίζονται καθόλου τα θέματα τη απασχόληση, τα θέματα τα κοινωνικά. Ήδη από τη συνθήκη μα έχει ζητηθεί αυτά τα εχέγγυα για την απασχόληση να τα συντονίζουμε μεταξύ μα. Κοινωνική προστασία, κοινωνική οικονομία ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει μία ανέλικτη ε, στρατηγική που επιβάλλει δημοσιονομικές πειθαρχίες, μία στρατηγική που δεν λειτουργήσε και που νομίζω ότι ε, είναι άλλωστε ε, και καταδικασμένη στην αποτυχία. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε. Η νομισματική ένωση όταν δεν συνοδεύεται από οικονομική και κοινωνική ένωση δεν είναι βιώσιμη. Και για το λόγο αυτό ζητήσαμε, όπως μας είπε και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να έχουμε μια κοινωνική διακυβέρνηση ε, στο ευρύτερο, με τον ευρύτερο ορισμό που θα αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και εκεί να έχουμε με πιο σφαιρική αντιμετώπιση, με κοινωνικές επενδύσεις που θα συνδέονται με τους στόχους της Ευρώπης 2020. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει η νομισματική ένωση. Είναι ένα μέσο ή είναι ένα στόχος. Ένα μέσο είναι η ευημερία για τους πολίτες μας. Χρειαζόμαστε ένα κοινωνικό πρωτόκολλο που θα εξασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα και μια δραστήρια πολιτική για την απασχόληση. Και θέλουμε να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ε, στηρίξει και η ίδια ε, την κοινοτική προσέγγιση και να μην κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα θίξουν τη θέση του Κοινοβουλίου. Και μια τελευταία παρατήρηση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευτεί περισσότερο για το εργαλείο αυτό, για το μέσο ε, το διατροφικό που θα εξασφαλίσει ε, τα εκατομμύρια συμπολιτών μας που αυτή τη στιγμή ζουν σε συνδίκες φτώχειας και πείνας. Και θα πρέπει αυτό να γίνει πάντα σε συνειδητονισμό και με τις εθνικές δικήσεις. Εκ μέρους του Άλντε, ο κύριος Νταφ. Κύριε Πρόεδρε. Ε, Πρόεδρε, ο κύριος Μπαρόζο έκανε λόγο για την δημοσίευση του σχεδίου του, του προτύπου του για όλα αυτά τα στοιχεία που θα χρειαστούμε και θα πρέπει να εφαρμοστούν για μια αυθεντική οικονομική και νομισματική ένωση. Δεν κατανόησα απόλυτα αν αυτού του είδους ε, οι κύβοι, τα στοιχεία θα συμπεριλάμβαναν ένα σχέδιο πρότασης για, την, για ένα ταμείο διάσωσης ε, και θα ήμουν ευγνώμων αν ο Επίτροπος Σεφτσοβιτς θα μπορούσε να το αποσαφηνίσει αυτό. Θα ήταν άκρος προβληματικό για το Ευρωκοινοβούλιο να συμφωνήσει για τα διπλά αυτά μέτρα για το 2-pack τη απουσία ωστόσο του Ταμείου Εξαγοράς Σωτηρίας. Δεύτερον, Redemption Fund. Δεύτερον, μετά από την ατυχή εξαφάνιση του πρώην Επιτρόπου Ντάλι ποια θα είναι η έκβαση τελική των καπνικών προϊόντων. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο και ο κύριος Σεφτσοβίτσε ελπίζω ότι θα είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει αυτή τη στιγμή, έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Τάλι και έτσι θα μπορούσε να μας ενημερώσει τι γίνεται με τα προϊόντα αυτά. Και επιπλέον Καλό το ότι υπάρχουν προσχέδια και προγράμματα για την ανάπτυξη της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι το πακέτο ως έχει για την νομοθεσία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς πόρο απέχει από το να είναι πλήρες. Η οδηγία περί παροχής υπηρεσιών που, έχει, που είναι κλειδί μέσα σε όλα αυτά δεν ε, υλοποιείται πλήρως ε, ακόμη σε διάφορα κράτη-μέλη, δεν εφαρμόζεται ακόμη. Και η οδηγία περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εξακολουθεί να εκκρεμεί και αναμένει ε, διευθέτηση, επίλυση. Και επίσης θα η επιθυμία του να τονιστεί η σημασία, η σπουδαιότητα των προγραμμάτων που τρέχουν τώρα και βρίσκονται σε εξέλιξη και πρέπει να υλοποιηθούν είναι δεδομένη για όσα εργαστήκαμε και θέλουμε να υπάρξουν και να λειτουργήσουν ως ρυθμίσεις και κανονιστικά προτού προχωρήσουμε περαιτέρω στην τελευταία φάση ας το έτσι των υψηπέδων των της φωτεινής διαδρομής προς την ενιαία εσωτερική αγορά που θα ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ. Και τώρα κυρία Ριβάζη για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή την εβδομάδα θα δώσουμε, ε, θα δώσουμε την απαλλαγή, τουλάχιστον θα ψηφίσουμε για την απαλλαγή κάποιων ευρωπαϊκών υπηρεσιών που είχαν πρόβλημα με τους προπολογισμού τους και θα δούμε μέχρι πού θα προωθήσουμε τη διαφάνεια για να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Την εβδομάδα αυτή που ζητήσαμε τα θεσμικά όργανα να είναι υποδειγματικά και να μην έχουν σύγκρουση συμφερόντων, τη στιγμή που για μια φορά ακόμα η φήμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατακυρώνεται, καταρακώνεται, με συγχωρείτε, εκ μέρου των Πρασίνων αλλά και πολλών άλλων Ευρωβουλευτών. Θέλω να σα ζητήσω τι γίνεται με το θέμα τη παρέτηση του κυρίου Ντάλι και με την αναθεώρηση τη οδηγία του για τα προϊόντα καπνού και καπνικών προϊόντων που εκκρεμεί εδώ και πάρα πολύ ε, καιρό. Πρέπει να σα πω πω τελώ σε σύγχυση. Γιατί υπάρχει κάτι ε, το εξαιρετικά ύποπτο πίσω από αυτή την ιστορία και έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε λεπτομέρειες. Βεβαίως, δεν είναι υπεράνω του νόμου οι επίτροποι. Βεβαίως πρέπει να λογοδοτήσουν όπως όλοι οι πολίτες μας. Αλλά οι επίτροποι δεν θα πρέπει να, είναι, να έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους υπόλοιπους. Και νομίζω ότι δεν δίνουμε ε, στον ε, ε, επίτροπο Ντάλι το δικαίωμα του τεκμηρίου της αθωότητας. Και θεωρούμε πως είναι ένοχος χωρίς να τον έχουμε ακούσει. Πολλά θέματα προκύπτουν και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας φωτίσει Ποιε είναι οι νομικές διατάξει, ποιο είναι ο κανονισμός ή η συνθήκη που παραβίασε ο κύριος Ντάλι με τη συμπεριφορά του. Τι θεωρεί πως συνέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ε, ένοχος ή πρόκειται για μια μανούβρα η οποία προσπαθεί να ε, σπρώξει στην άκρη αυτή την οδηγία για τον καπνό και τα καπνικά προϊόντα. Θα ήθελα κύριε Επίτροπε να μας δώσετε διευκρινήσεις για αυτή την έκτακτη περίσταση και νομίζω ότι θα πρέπει και η Όλαφ να μας στείλει την έκθεσή της το συντομότερο δυνατόν. Διάβασα το, το mail που έστειλε ο κύριος Μπαρόσο που μας είπε πως η οδηγία για τα προϊόντα καπνού δεν θα καθυστερήσει. Θέλουμε όμως να δούμε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα, γιατί ήδη καθυστερεί πάνω από ένα χρόνο. Η οδηγία είναι έτοιμη και σας ζητώ, ζητώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί για να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο αυτή η πολυανομενόμενη οδηγία για να δούμε τι θα συμβεί, γιατί σε επίπεδο υγείας πιέζει το θέμα, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσει να τρέχει αυτή η οδηγία, γιατί αν δεν γίνει τώρα θα περιμένει την επόμενη η θητεία, άρα λοιπόν θα έχει κερδίσει το λόμπι του καπνού. Ευχαριστώ κυρία Ριβάζη. Εκ μέρους της CCR ο κύριος Χάρμπουρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ομάδας μου και ε, όντα ένα από αυτού που εργάστηκαν για αυτό το πρόγραμμα και ω πρόεδρο ε, τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την, για την ε, εσωτερική αγορά, καλωσορίζω αυτέ τι προτάσει. Δεν υπάρχει τίποτα απροσδόκητο εκεί, αλλά θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σχετικά. Διότι θέλω να πω στον κύριο Σεύκοβιτ, δεν είναι αυτό καθόλου ουσιαστικά το πρόγραμμα εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα κατάλογο νέων πρωτοβουλειών. Και όπω είπαν πολλοί συνάδελφοι, Μπορεί να είναι σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες, αλλά έχει και τη σπουδαιότητά, τους, τη σπουδαιότητά της η εφαρμογή των προγραμμάτων που τρέχουν και έχουν ήδη δρομολογηθεί και υλοποιούνται. Και είναι πολύ σημαντικό, και εδώ υποστηρίζω αυτό το οποίο αρκετοί συνάδελφοι προανέφεραν ήδη, η υλοποίηση και εφαρμογή και η συμμόρφωση με τους υφιστάμενους κανονισμούς και οδηγίες είναι σημαντική υπόθεση. Για παράδειγμα για τον τομέα που γνωρίζω καλύτερα. Θα ολοκληρώσουμε του χρόνου και θα ολοκληρωθεί η οδηγία περί δημοσίων προμηθειών. Και αυτό θα απαιτήσει ευρύτατη εφαρμογή και κατάρτιση στα κράτη-μέλη για να είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα. Θέλω να πω το εξή προ εμά, κύριε Σεύτσοβιτ. Στο μέλλον, το έργο σα πρέπει να είναι το πλήρε ε, πρόγραμμα εργασιών ε, Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και θέλουμε να δούμε ποια πρόοδος θα έχει επιτευχθεί σε σχέση με όλου αυτού του τομεί. διότι αυτό έχει κέρια σπουδαιότητα θέλουμε να δούμε αυτά τα προγράμματα θέλουμε να δούμε τι θα πράτεται σχετικά και ο συνάδελφος Άντριου Ντάφ ανέφερε την οδηγία περί υπηρεσιών που η δική μου κοινοβουλευτική επιτροπή δραστήρια παρακολουθεί και εργάζεται επ' αυτή. και εδώ πάλι έχουμε ένα κατάλογο των ιδεών σας ε, τι μπορεί να απλουστευτεί και τι μπορεί να επιτευχθεί με αυτόν τον οργανισμό. Θέλω να σα υπενθυμίσω στο πρόγραμμα εργασίας μας υπάρχει και το ψήφισμα το οποίο σχολιάστηκε. Συγκεκριμένα ζητήσαμε εκεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιωθεί η ποιότητα του νομοθετικού σχεδιασμού και να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει η αξιολόγηση επιπτώσεων και όλων αυτών των συναφών. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα από όλα αυτά. Γιατί και γνωρίζουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής εργάζεται επί αναθεωρήσεως αυτών, πάλι Ούτε λέξη δεν ε, αναφέρθηκε επ' αυτού την επιφορά. Να μας αποστείλετε παρακαλώ το πρόγραμμα εργασίας πρωτοβουλειών ποιότητας, ε, ποιοτικών δράσεων και εφαρμογής, υλοποίησης. Να το κάνουμε αυτό πλήρως ε, κύριε Σεφτσοβίτση και όχι επιλεκτικά και να μην έχουμε εδώ κάποιες νέες πρωτοβουλίες και τελεία και παύλα. Ας κάνουμε το πλήρες έργο όπως απαιτείται και καλύτερα. Η κυρία Άντερσον έχει το λόγο για τους για την Πολλά είναι σωστά στο πρόγραμμα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά τα προβλήματα κρύβονται στις ε, δυσκολίες και αναφερθήκατε εσείς σε 7 τομείς πολιτικής. Εκεί θέλουμε εμείς να κάνουμε μια ε, συμβολή επικοδομητική για να δούμε πώς μπορούμε να ωφελήσουμε τους Ευρωπαίους γενικότερα. Για το πρόγραμμα λοιπόν θεωρούμε πως πρόκειται για μια ακόμα χαμένη ευκαιρία. Θέλουμε μια ριζικά τροποποιημένη προσέγγιση. Δεν αναφερθήκατε καθόλου στι οδηγίε για τον καπνό και τα καπνικά προϊόντα που καθυστερούν εδώ και καιρό και χρειάζεται οι ανάγκε των ατόμων να υπερισχύσουν των οικονομικών ο, Υπάρχει λοιπόν νομοθεσία η οποία θίγει ιδιαίτερα τα παιδιά και τις γυναίκες. Οι δημοσιονομικές περικοπές, για παράδειγμα, αύξησαν τα ποσοστά φτώχειας σε παιδιά, σε γυναίκες και για την ανάπτυξη και την απασχόληση δύσκολα βρέπει κανείς να υπάρχουν μέτρα που θα προωθήσουν την απασχόληση και νομίζω ότι δεν χρηματοδοτούνται αρκετά. Έχετε κάποια ιδεολογική προσκόλληση στις δημοσιονομικές, στα δημοσιονομικά μέτρα πειθαρχίας του ελλείμματος και βλέπετε πως οι επιδόσεις δεν είναι θετικές παρόλα αυτά. Είναι απογοητευτικό που εσείς δεν αναφέρεστε καθόλου στις αποτυχημένες πολιτικές που προσπαθούν να επιβάλλουν όρους τρίτου κόσμου στην απασχόληση, στις υπηρεσίες που ε, προσφέρονται. Με το να ρίχνουμε τους μισθούς και να καταστρέφουμε τις ε, θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να κερδίσουν δισεκατομμύρια λίρες οι τράπεζες. Και μετά τα όσα είπε το Σεπτέμβριο για την κατάσταση της Ένωσης ο πρόεδρος κ. Μπαρόσα είπα πως νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να ε, ε, αλλάξει νοτροπία. Και ελπίζω να το κάνετε και εσείς κύριε Αντιπρόεδρε και να καταλάβετε τι βλάβη έχετε προκαλέσει στη ζωή του κόσμου με αυτά τα ε, μέτρα λιτότητας που έχετε επιβάλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Άντερσον και σας ευχαριστώ που ήσασταν η μοναδική μάλλον η οποία σεβάστηκε τους χρονικούς περιορισμούς. Ο κύριος Σιμάνσκι έχει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την πρόθεση μεταξύ άλλων την υλοποίηση, την εφαρμογή του προγράμματος ε, για τις κλιματικές ε, αλλαγές. Το 2013 είναι το έτος όπου θα περάσουμε στην τρίτη φάση του ETS, του συστήματος εμπορίας ρήπων. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο και περισσότερο ασχολείται με τα δικαιώματα παρέμβασης ε, στις οικονομίες. Ούτε το Κοινοβούλιο ούτε τα κρατη θα έπρεπε να εγκρίνουν αυτή τη δράση. Το πρόγραμμα, το σχέδιο για τις εκπομπές ρήπων και για την μείωση των εκπομπών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα είναι μόνο ένα παράδειγμα της παρεμβατικής δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορεί να οδηγήσει στην κρίση αυτή οι οικονομίες μας να υποστούν ακόμα μεγαλύτερη ένταση και πίεση και αυτό φυσικά ε, να δούμε και το τι γίνεται για τις οικονομίες που εξαρτώνται από το ε, λιθάνθρακα και γι' αυτό πιστεύω ότι η τροπολογία ή το αίτημα των δικών μου ε, συμπολιτών σε σχέση με το πακέτο αυτό για τις κλιματικές αλλαγές θα έπρεπε λοιπόν να πάψει να ισχύει διότι έχει αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό θέλουμε να ζητήσουμε και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Πριν από ένα χρόνο, πριν από ένα έτος, ε, ανακήρυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έτος των πολιτών. Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν έχουν σαν στόχο την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των λαών την Ευρώπη. Ήφεση, ανεργία, υποαπασχόληση, μειωμένες ε, κοινωνικές παροχές και τα μέτρα οστέρησης έχουν, ε, λιτότητας έχουν ακριβώς σαν στόχο την αύξηση αυτής της λιτότητας και την ύφεση. Η Ευρώπη λοιπόν αντιπροσωπεύει κάτι το οποίο δυστυχώς έχουν υπερεκτιμήσει ιδιαίτερα οι λαοί του Νότου οι οποίοι υποφέρουν από την ε, οικονομική ύφεση. Άλλη πρόταση είναι να χρησιμοποιηθούν πόροι της Ένωσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Οι χώρες οι οποίες δεν έχουν υποτιμημένα νομίσματα όμως δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα πρέπει να ανταγωνιστούν τις βιομηχανίες από τις χώρες τις αναπτυσσόμενες με απαράδεκτες συνθήκες παραγωγής. Αντιπρόεδρος κ. Σεύκοβιτς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στα περισσότερα σχόλια. Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να σας δώσω ένα έγγραφο γιατί το τελικό πρόγραμμα υιοθετήθηκε εδώ και μια μισή ώρα και μου ζητήθηκε να σας το παρουσιάσω αμέσως άμα τη αποδοχή του. Θα είναι όμως σύντομα διαθέσιμο σε όλους σας και θα, σήμερα το απόγευμα. Σχετικά με την σχέση ανάμεσα στις κατεξουσιοδότηση πράξεις και τις εφαρμοστικές πράξεις. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο πότε θα χρησιμοποιούμε τα μεν και πότε τα δε. Η πηγή των προτάσεων μας ανάλογα με το είδος των προτάσεων είναι κάτι που καθορίζεται από τη συνθήκη είναι σαφές για ποιες πολιτικές απαιτούνται εφαρμοστικές πράξεις και για ποιες πολιτικές απαιτούνται κατεξουσιοδότηση πράξεις. Αυτό το συζητήσαμε και με τη διάσκεψη των Προέδρων και με τη διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επίτροπων. Απαιτείται να συντονίσουμε καλύτερα την νομοθετική μας διαδικασία γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει συχνά είναι ότι η αντίθεση ανάμεσα στα δύο είδη ε, πράξεων γίνεται ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα πλαίσια της διαδικασίας, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, κάτι το οποίο δεν είναι απολύτως νόμιμο και γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε από το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, <clears throat> θα ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τελικά η ανατροπή κάποιων αποφάσεων οι οποίες έχουν ληφθεί αν ακολουθήσουν την άποψη των μεν ή των δε. Θα πρέπει λοιπόν να σεβόμεθα τη συνθήκη και να μην χρησιμοποιούμε σαν διαπραγματευτικό χαρτί της κατεξουσιοδότηση πράξεις και τις εφαρμοστικές πράξεις. Απαιτείται να μειώσουμε την περιπλοκότητα και τη γραφειοκρατία. Υπάρχουν προτάσεις για τη μείωση του λεγόμενου διοικητικού άχθους κατά 31% και θα προσπαθήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε τις βελτιώσεις αυτές πώς μπορούμε να τις κάνουμε πραγματικότητα στα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί ναι μεν συνεργαζόμαστε σωστά με τα κράτη-μέλη, αλλά δεν βλέπουμε και δεν ελέγχουμε αν οι απλουστεύσεις τις οποίες εμείς επιτυγχάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πηγαίνουν ε, στις ε, χώρες μέλη. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Χάρμπορ ότι πάντα υπάρχει δυνατότητα βελτίωση σε σχέση με τις μελέτες επιπτώσεων. Κάνουμε προσπάθεια εδώ και αρκετό καιρό. Χαίρομαι που και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να κάνει και αυτό τέτοιου είδους μελέτες για τροπολογίες τις οποίες αυτό προτείνει και νομίζω ότι μέσα από αμοιβέ προσπάθειες θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις προτάσεις μας σχετικά τώρα με την αποδοτικότητά μας. Για το 2020 έχει υπάρξει πρωτοβουλία για 16 πρωτοβουλίες. Είμαστε στις 8 πριν από το τέλος του χρόνου. Νομίζω ότι αν δεχθούμε ε, τις παραδοσιακές θα έλεγα μορφές εκτέλεσης των προγραμμάτων είδαμε ότι το 2010 και το 2011 είχαμε φτάσει στο 90% του συνόλου των προγραμμάτων τα οποία είχαμε προαναγγείλει στην προηγούμενη περίοδο. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα να φανούμε αποδοτικοί εδώ. Σχετικά με την κρίση της ε, απασχόλησης, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό είναι βασική μας προτεραιότητα. Και από τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις νομίζω ότι το κατανοήσατε αυτό. Ήδη από τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο μάλλον θα κάνουμε προτάσεις για την απασχόληση των νέων για τις εγγυήσει για την απασχόληση των νέων και επί τη βάση της εμπειρίας της οποίας είχαμε μέχρι τώρα και μέσω των ομάδων δράσης που στείλαμε στις χώρες όπου υπάρχει υψηλότατο επίπεδο ανεργίας των νέων. Η σωστή και γρήγορη χρήση των ταμείων μπορεί να δημιουργήσει 400.000 θέσεις απασχόλησης Σήμερα το πρωί μιλήσαμε και για το πολιετές πλαίσιο υπάρχει μια γραμμή η οποία επαναλαμβάνεται σε όλες τις ομιλίες μου και τις παρατηρήσεις μου. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το 25% των κοινοτικών ταμείων στα πλαίσια των μελλοντικών προοπτικών έχουν σαν στόχο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η Επιτροπή είναι ξεκάθαρο. Λέμε ότι η αδίποτε μείωση του ποσοστού αυτού είναι απαράδεκτη για την Επιτροπή. Και ελπίζω να είμαστε ικανοί να πείσουμε τα κράτη-μέλη γι' αυτό γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι ο καθρέφτης αν θέλετε της προσπάθειας την οποία κάνουμε χρησιμοποιώντας τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη τύχη στην απασχόληση οι πολίτες της Ένωσης. Ένα τελευταίο θέμα ήταν η κατάσταση σχετική με τον προηγούμενο επίτροπο, τον συνάδελφο, τον κύριο Ντάλι και την οδηγία για τα προϊόντα καπνού σχετικά με την παρέτηση του Επιτρόπου κυρίου Ντάλι. Ήταν σαφές ότι μετά από την έρευνα της ΟΛΑΦ και μετά από τη συζήτηση της έκθεσης της ΟΛΑΦ ανάμεσα στον πρόεδρο της Επιτροπής και τον Επίτροπο ήταν σαφές ότι η θέση του ήταν πάρα πολύ δύσκολα, ήταν ανυπόφορη θα έλεγα σε σχέση με την φήμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη δική του. Γι' αυτό λοιπόν Ξεκινήσαμε τη διαδικασία για το διορισμό του νέου Επιτρόπου. Νομίζω ότι και μετά από τις πρώτες επαφές που είχα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουμε την ακρόαση του νέου Επιτρόπου μέσα σε λίγες εβδομάδες και ο νέος Επίτροπος θα μπορέσει να αναλάβει το ταχύτερο δυνατόν. Ήδη συζήτησα το πρόγραμμα για τις επόμενες εβδομάδες με τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Θα έχουμε και τη συνάντηση με τον κύριο Χάρμπορ σε λίγη ώρα και θέλω να είμαι σίγουρος ότι η προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει θα συνεχιστεί. Όλες οι διαδικασίες τριμερούς διαλόγου θα συνεχιστούν και για τα προϊόντα καπνού είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για την οδηγία προϊόντων καπνού. Να παρουσιάσουμε μια καλή πρόταση πάνω στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει τουλάχιστον την πρώτη ανάγνωση. Θα ήταν βέβαια σωστότερο να μπορούσε ο νέος Επίτροπος να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή εξ αρχής, από την αρχή μέχρι το τέλος, στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου αλλά νομίζω ότι βλέποντας το χρονοδιάγραμμα για τον διορισμό του νέου Επιτρόπου ότι δεν θα καθυστερήσουμε. Είναι λοιπόν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει την οδηγία για τα προϊόντα καπνού εγκαίρως και να αποφασίσετε από εκεί και πέρα εσείς. Ευχαριστώ κύριε Στευκόβιτς. Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013 ολοκληρώθηκε και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η σύσταση του κυρίου Μορέιρα πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ευρωπαϊκής κοινότητας